κυρία Κρόνπερ, για 1,5 λεπτό μεταξύ των συντακτών της, ε, του θέματος, του ψηφίσματος. Ευχαριστώ. Πρόσφατα πάρα πολύ έχασαν τη ζωή τους έξω από την πρωτεύουσα του Μπαγκλαδέ, σύμφωνα με την αστυνομία. 18 έχασαν τη ζωή τους, σκοτώθηκαν, λέει η έκθεση. Πρέπει λοιπόν να προβούμε σε έρευνες με διαφάνεια και αντικειμενικές για να διευκρινιστούν τέτοιες και άλλες περιπτώσεις. Μα ανησυχεί ιδιαίτερα η συνεχιζόμενη βία και η παράλυση βασικά του κράτου του Πακλαντέ και η αντιπαράθεση που υπάρχει μεταξύ των δύο πολιτικών πλευρών. Είναι θλιβερό που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα πολιτικά κόμματα δεν καταφέρουν να καταλήξουν σε ένα συμβασμό τόσο αναγκαίο προκειμένου οι κάτοικοι του Μπαγκλαντές να μπορέσουν να εκφράσουν τη βούλησή τους για πολιτικές αλλαγές. Η κατάσταση χειροτερεύει. Το Μπαγκλαντές προσπαθεί να ανακάμψει από την φτώχεια και να αναδιορθώσει τη βιομηχανία του. Όμως έγιναν οι καταστροφές, ε, Κρεμίστηκε το εργοστάσιο όπως ξέρουμε, με 1.100 εργαζόμενους, οι συνθήκες εργασίας είναι πάρα πολύ σκληρές, εκεί που απασχολούνται 4 εκατομμύρια άνθρωποι. Κάνουμε λοιπόν έκκληση και ζητάμε ε, σε όλες τις πλευρές στη χώρα να μην υπονομεύσουν ακόμα περισσότερο την υπόλοιπη ε, πολιτική και οικονομική σταθερότητα του Μπαγκλαντές. Ο λόγο του Μπαγκλαντές χρειάζεται χρήματα. Ευχαριστώ. Ευχαριστή, ευχαριστώ. Ο κύριος Κόβαλ για ένα λεπτό ακολουθεί. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Τα γεγονότα των τελευταίων εβδομάδων στο Μπαγκλαντές έχουν οδηγήσει σε μεγάλη απογοήτευση από τη δική μας πλευρά. Ελπίζουμε, ελπίζαμε ότι η εκλογή θα ήταν μια ευκαιρία για να μπορέσει να λειτουργήσει η ειρηνική αλλαγή στο πολιτικό στερέωμα. Αυτό όμως δεν έγινε. Το ψήφισμά μας είναι μια απάντηση σε αυτή την κατάσταση και είναι και αποτέλεσμα του ενδιαφέροντος που έχουμε για τον Μπαγκλαντές. Και ο λαός του Μπαγκλαντές περιμένει να ακούσει ποια είναι η θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για ένα σημαντικό θέμα δεν είναι μόνο ένα πολιτικό θέμα, αλλά είναι και θέμα θρησκευτικό. Μας ενοχλεί και μας απασχολεί το θέμα ότι υπήρξαν επιθέσεις κατά των χριστιανών τις ημέρες των εκλογών. Θα πρέπει να δώσουμε ένα σαφές μήνυμα ότι μας ενδιαφέρει και θέλουμε να υποστηρίξουμε τις δυνάμεις αυτές οι οποίες θέλουν να εισαγάγουν μια πιο ειρηνική κατάσταση στο Μπαγκλαντές και θα πρέπει να υπάρχει μια ελάχιστη τουλάχιστον συμφωνία μεταξύ των πολιτικών δυνάμεων στον Παγκλαντέ. Ευχαριστώ κύριε Κόβαλ. Η κυρία Ντεκέζερ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αμφιλεγόμενες εκλογές έγιναν στο Μπαγκλαντές, οι οποίες οδήγησαν σε κλιμάκωση της βίας με 21 τουλάχιστον θύματα. Δεν είναι σαφής οι αριθμοί, αλλάζουν σύμφωνα, αλλά σύμφωνα με τις ε, πηγές ε, είναι μια χώρα ε, η οποία, ε, μια φίλη χώρα ε, η οποία έχει πληγεί από πολλές τραγωδίες που συζητήθηκαν εδώ. Πρέπει να σας πούμε ότι εδώ στις προκείμενες εκλογές είχαμε μποϊκοτάζ από πλευρά του Εθνικιστικού ε, Κόμματος του ε, Μπαγκλαντές που στις προηγούμενες εκλογές ε, είχε πάρει 45% το 2001 και 2 τρίτα των εδρών στην Βουλή. Επομένως το μποϊκοτάζ αυτό τροποποίησε πάρα πολύ τις εκλογές οι οποίες είδαν ένα πάρα πολύ μικρό ποσοστό ε, συμμετοχής ε, με αποτέλεσμα ε, τα αποτελέσματα, η έκβαση των εκλογών να είναι ιδιαίτερα εύθραυστη ζητούμε ενδεχομένως να γίνουν νέες εκλογές αν αυτό είναι απαραίτητο. Ευχαριστούμε κύριε Ντεκάζερ και ως Μπένιον για 1,5 λεπτό. Μπορώ να ξεκινήσω, βεβαίως. Σα ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και εγώ λυπάμαι πάρα πολύ για το γεγονό ότι το Μπαγκλαντέ δεν μπόρεσε να έχει μια περιεκτική και δημοκρατική διαδικασία εκλογών. Εμεί πιστεύουμε σε μια ελεύθερη κοινωνία όπου ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράσει την άποψή του και αυτό αποτελεί αναγκαιότητα να υπάρχουν αξιόπιστε και ελεύθερε εκλογέ. Και η κυβέρνηση και οι αντιπολίτευση του Αγγλαντές θα πρέπει να θέσουν πρώτο το συμφέρον του λαού του Μπαγκλαντές και να βρουν μια συμφωνία, μια φόρμουλα για να υπάρξει η δυνατότητα να ξαναγίνουν οι εκλογές το ταχύτερο δυνατόν. Να υπάρξει μια συμβαστική λύση που θα δώσει και πάλι τη φωνή τους στους πολίτες του Μπαγκλαντές και θα σεβαστεί αυτή τη φωνή. Εγώ Λυπάμαι για τη βία που χρησιμοποιήθηκε για να μην ψηφίσουν οι πολίτες αλλά και την αυθαίρετη κράτηση των πολιτικών της αντιπολίτευσης που πρέπει να απελευθερωθούν. Δεν ε, εξέρω ιδιαίτερα το ρόλο του ε, Δικαστηρίου Διεθνών Εγκλημάτων που οδήγησε σε πόλωση της ε, κοινωνίας του Μπαγκλαντές, χρησιμοποίησε την θανατική ποινή με καταχρηστικό τρόπο και έχει οδηγήσει σε περαιτέρω διχασμό στον Μπαγκλαντές. Και με εκπλήσει και με αποτροπή πιάζει ότι το Βρετανικό Συντηρητικό Κόμμα, οι Τόρις, υποστηρίζουν την εφαρμογή του, της θανατικής ποινής στο Μπαγκλαντές και παροτρύνω την ύπατη εκπρόσωπο την κυρία Άσο να ασκήσει διπλωματική πίεση για να μπορέσει να υπάρξει μια λύση. Αυτή ήταν και η ελπίδα που είχαμε ε, μετά από τη δήλωση του ηγέτη της αντιπολίτευσης σήμερα το πρωί που είπε ότι η αντιπολίτευση θα σταματήσει τις διαμαρτυρίες και τις διαδηλώσεις και θα προσπαθήσει να υπάρξει μια συμβαστική λύση. Ας ελπίσουμε ότι αυτό θα γίνει για να μπορέσουμε να σεβαστούμε τις θεμελιώδεις ελευθερίες των Παγκλαντές. Ευχαριστώ κύριε Μπένιον. Ο κύριος Τάνοκ για διαδικαστικό θέμα. Το, αναφέρθηκε το συντηρητικό κόμμα από τους ε, φιλελεύθερους από το Ηνωμένο Βασίλειο. Πρέπει να σας πω ότι το συντηρητικό κόμμα θεωρεί ότι είναι θέμα συνείδησης για τον καθένα. Δεν έχουμε ε, ως κόμμα άποψη σχετικά με την θανατική ποινή. Είναι θέμα συνείδησης του καθενός. Ευχαριστούμε για 1,5 λεπτό η κυρία Σόσα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αναφέρθηκαν ήδη τα γεγονότα τα οποία στιγμάτισαν τις πρόσφατες εκλογές του Μπαγκλαντές και η κλιμάκωση βίας που ακολούθησε και οδήγησε στο θάνατο πολλών ατόμων. Και επίσης η φυλάξη πολλών πολιτικών ηγετών της αντιπολίτευσης. Είναι απαραίτητο να υπάρξει μια ανεξάρτητη επιτροπή έρευνας η οποία να μπορέσει να διαπιστώσει τι ακριβώς έγινε αλλά επίσης να απελευθερωθούν οι κρατούμενοι. Είναι μια κατάσταση λοιπόν που έχει χαρακτηριστεί από βία καταστολή πολλών απεργιών και διαδηλώσεων. Το Μπαγκλαντές είναι μια χώρα όπου οι συνθήκες εργασίας είναι άθλιες. Υπάρχει μια εκμετάλλευση χωρίς όρια των εργαζομένων και θυμόμαστε όλοι ότι είχαμε συζητήσει πρόσφατα την, ε, το πρόσφατο ψήφισμα για την κατάρρευση ενός εργοστασίου κλωστοεφαντοργικών που οδήγησε στο θάνατο χιλίων και περαιτέρω ανθρώπων. Πρέπει να τονίσω επίσης ότι είναι απαραίτητο τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να έχουν το θάρρος να εξαλείψουν από τις δημόσιες προμήθειές τους τι εταιρείε οι οποίες έχουν εργαζομένου σε τέτοιες συνθήκες στον Παγκλαντέ. Ευχαριστώ κυρία Σόσα. Ο κύριος Κάσμαρεκ για ένα λεπτό έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Στην αρχή του 2013 σκοτώθηκαν πάνω από 3.000 άνθρωποι ε, στο Πακιστάν, 18 εκ των οποίων την ημέρα των εκλογών οικονομική και κοινωνική πρόοδος ε, που επετεύχθη μέχρι τώρα στην, ε, στο Μπαγκλαντές οπωσδήποτε απειλείται από αυτήν την ε, βία. Η θανατική ποινή επίσης είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό ζήτημα. Μία πάυση, ένα μορατόριουμ στις θανατικές ποινές θα μπορούσε να ελαφρύνει λίγο την κατάσταση τα, ε, κράτη, τα ε, πολιτικά κόμματα θα πρέπει να σταματήσουν την βία καθώς επίσης και οποιαδήποτε μορφή ε, επίθεσης και βίας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Αυτά ήταν αυτές ήταν οι ομιλήσεις από τους συντάκτες. Τώρα αρχίζουν οι ομιλητές εξωρώματος πολιτικών ομάδων με τον κύριο Πόσελ για ένα λεπτό πρώτα. Κύριε Πρόεδρε. όταν ήμουν εγώ νέος θυμάμαι τον πόλεμο της ανεξαρτησίας του Πακιστάν, του Μπαγκλαντές, συγγνώμη. Την διάλυση του Πακιστάν και τα δραματικά αυτά γεγονότα τα οποία λαμβάναν χώρα την εποχή του πολέμου της Ινδοκίνας. Υπήρξαν κάποιες δυναστείες οι οποίες έχουν έκτοτε ε, λαιλατήσει και κυριαρχήσει στο Μπάγκλαντες που έχουν καταδικάσει τον πληθυσμό σε φυσικές καταστροφές και ακραία ένδια. Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει δυνατόν να επιτευχθεί μια σχετική ευμάρεια στη χώρα αυτή και να ανοίξει ο δρόμος του μέλλοντος για τον Μπαγκλαντές. Αλλά αυτός ο δρόμος δεν θα μπορέσει να προχωρήσει παρά μόνο όταν βασίζεται στη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα και όχι στην προπαγάνδα. Θα πρέπει να τηρήσει τις δημοκρατικές αρχές και στον εμπορικό και οικονομικό τομέα. Δεν μπορεί να βασίζεται στην ε, φθηνή εργασία σε εργοστάσια, φυλακέ, αλλά είναι απαραίτητο να υπάρξει δημοκρατία στον Μπαγκλαντέ. Ευχαριστώ πολύ. Ακολουθεί για ένα λεπτό ο κύριος Ρέπο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Οι κοινοβουλευτικές εκλογές στο Μπαγκλαντές ήταν δυστυχώς αποτυχία εξαιτία της βίας. Το 2013 ήταν η χρονιά η πιο καταστροφική από την ανεξαρτησία της χώρας και μετά. Εδώ έχουμε τις θέσεις των δύο αντίθετων κομμάτων που περιπλέκει την κατάσταση ακόμα περισσότερο. Επίσης, υπάρχουν και επιθέσεις κατά των πολιτιστικών και θρησκευτικών μειονοτήτων. Πρέπει λοιπόν να γίνει έρευνα μετά από τον θάνατο που προκάλεσε και τον άτους μάλλον που προκάλεσε η πανέβαση των αστυνομικών αρχών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν πρέπει να φροντίσει να υπάρξει ειρηνική κατάσταση εκεί και να μην επιτρέπεται πια θανατική ποινή. Υποφέρει ο λαός εκεί και αν δεν υπάρξει η εθνική συμφιλίωση η χώρα δεν θα μπορέσει να πάει μπροστά. Ευχαριστώ. Ε, το λόγο. Οι εκλογές ε, στο Μπαγκλαντές ε, κατέδειξαν ότι η χώρα έχει προβλήματα δημοκρατίας ε, ε, και πρέπει να τα αντιμετωπίσει. Η δράση του Διεθνούς Δικαστηρίου αποτέλεσε ε, την σωστή το σωστό τρόπο αντιμετώπισης, έστω και αν η αντιπολίτευση προσπάθησε να υπονομεύσει τη δράση του δικαστηρίου. Η εμπειρία της ε, τελευταίας υπηρεσιακής ε, κυβέρνησης ε, έδειξε ότι ήταν σωστή η προσέγγιση, ήταν σωστός ο τρόπος με τον οποίο προσέγγισε τις καταστάσεις. Ελπίζω ότι η νεοεκλεγήσα κυβέρνηση θα μπορέσει να λύσει ορισμένα από τα προβλήματα που προκλήθηκαν από μια ανεύθυνη αντιπολίτευση. Ευχαριστώ κύριε Τσανέσκι. Για ένα λεπτό ο Πάσκα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Οι αντιπαραθέσεις μεταξύ της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης στο Μπαγκλαντές έχει οδηγήσει σε μια κλιμάκωση της βίας και το γεγονός ότι το Εθνικιστικό Κόμμα του Μπαγκλαντές που είχε μποϊκοτάρει τις εκλογές μαζί με τη, τη χαμηλή προσέλευση στις εκλογές έχει υπονομεύσει την ε, νομιμοποίηση της νίκης της Λίγας Σαγουάμι. Για αυτούς τους λόγους θα πρέπει να δημιουργήσουμε τις απαραίτητες προϋποθέσεις ώστε να προχωρήσει ο διάλογος των πολιτικών δυνάμεων, ώστε να μην υπάρξει περαιτέρω κλιμάκωση και όξυνση της βίας. Μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορεί να προχωρήσει μια διαδικασία δημοκρατίας μέσω μιας ε, υπηρεσιακής κυβέρνησης ή με, μέχρι την επανάληψη των εκλογών και χωρίς ε, αντίπεινα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πάσκα. Ο κύριος Κούκαν για ένα λεπτό πάλι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η κατάσταση στο Μπαγκλαντές είναι κρίσιμη. Κάποια προβλήματα δεν είναι καινούρια στο Μπαγκλαντές, αλλά υπάρχει μια όξυνση της βίας μετά από τις εκλογές. Θέλω να κάνω μια έκκληση στην κυβέρνηση του Μπαγκλαντές να κάνει σαφή, να αναλάβει σαφή ευθύνη για τις διεθνείς υποχρέωσεις και να σταματήσει η βία δράση της αστυνομίας εναντίον γυναικών και παιδιών. Όλα αυτά δεν μπορούν να θεωρηθούν ότι είναι αποδεκτά και ο θάνατος των 18 α, θυμάτων το συγκρούσεων με την αστυνομία θα πρέπει να τύχει διαλεύκανση, να πρέπει να υπάρξει και μια έκκληση σε διάλογο μαζί με την αντιπολίτευση. <clears throat> πρέπει να εξασφαλίσει η δημοκρατικοποίηση της κοινωνίας των Μπαγκλαντές με τη συμμετοχή όλων των πολιτικών δυνάμεων και την εθνική συμφιλίωση που είναι προϋπόθεση για μια λειτουργούσα δημοκρατία για πρώτη φορά μετά από το 1990 δεν εκπροσωπείται η αντιπολίτευση στο Κοινοβούλιο του Μπαγκλαντές. Αυτό δεν είναι κάτι το οποίο προωθεί την δημοκρατία ούτε αντανακλά τα αισθήματα του πληθυσμού. Ακολουθεί κυρία Αντρίκενα. Το Δεκέμβριο που μας πέρασε το ΕΛΚΑ υπό τη δικιά μου την ηγεσία οργάνωσε ακρόαση σχετικά με ελεύθερες εκλογές στον Μπακλαντές. Ήρθαν διάφοροι εκπρόσωποι και σήμερα όλοι γνωρίζουμε ποιο είναι το αποτέλεσμα των εκλογών εκεί και της κατάστασης που επικράτησε μετά τις εκλογές. Κάνουμε έκκληση λοιπόν στην κυβέρνηση της χώρας να σταματήσει όλα τα κατασταλτικά μέτρα από πλευρά τη αστυνομία και να ελευθερώσει όσου αυθαίρετα συνελήφθησαν από την αντιπολίτευση. Για να βγούμε από την πολιτική κρίση πιστεύω ότι πρέπει να σκεφτούμε όλε τι δυνατέ λύσει και ξανά με όλα τα νόμιμα πολιτικά κόμματα ώστε να μπορέσει ο κόσμος να επιλέξει. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα που έχει στη διάθεσή της για να βοηθήσει μια τέτοια διαδικασία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Αντρικένη. Ερχόμαστε στη διαδικασία ΚΑΣΤΙΑ. Σχεδόν 10 ομιλητές έχω που θέλουν να λάβουν το λόγο. Εγώ προέβλεπα μόναχα ένα ή δύο. Δυστυχώς δεν μπορώ να δώσω σε όλους το λόγο. Και ιδίω σε αυτούς οι οποίοι έχουν ήδη λάβει το λόγο. Κύριε Ίγκμα, έχει το λόγο πρώτα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Οι εκλογές που έλαβαν χώρα στο Μπαγκλαντές στην ουσία αρνούνται οποιαδήποτε αρχή δημοκρατίας όχι μόνο ε, ε, ε, σε σχέση με, την, με, με τους όρους αλλά και γιατί δεν υπήρξαν και ξένοι παρατηρητές η κατάσταση αυτή εκφράζει πραγματικά, ε, μάλλον η, έκβαση των εκλογών στην ουσία δείχνει την μεγάλη δυσαρέσκεια των ε, ε, εκλογέων. Άλλωστε είναι γνωστό ότι πολλά εκλογικά κέντρα αναγκάστηκαν να κλείσουν λόγω εμπρισμών η ε, αντιπολίτευση η οποία μποϊκοτάρισε τις εκλογές συνεχίζει να καλεί σε βία. Ε, θα πρέπει να σταματήσει η αιματοχυσία. Θα πρέπει να βρεθούν λύσεις. Ευχαριστώ πολύ. Σας παρακαλώ, να κλείσετε. Λέει ο πρόεδρος. Η κυρία Ευχαριστώ. Πάλι συζητάμε για το Μπαγκλαντές. Πριν από δύο μήνες είχαμε συζητήσει τη βία στον Παγκλαντές. Οι εκλογές του Ιανουαρίου που μποϊκόταρη αντιπολίτευση έκαναν το πρόβλημα ακόμα πιο μεγάλο στη χώρα. Η εξέγερση πριν τις εκλογές είχε σαν αποτέλεσμα 300 θύματα. Καταστράφηκε η διοκτησία. Και αυτό το οποίο είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό είναι ότι δεν γίνονται προσπάθειες για πολιτική συμφιλίωση και συμφωνία. Παρά την στήριξη που υπάρχει από τη διεθνή κοινότητα. Οι αρχές λοιπόν πρέπει να σταματήσουν τη βία κατά της αντιπολίτευσης, να σταματήσουν τις συλλήψεις, τους βασανισμούς και τις επιθέσεις σε βάρος των μειονετήτων. Ζητάμε επίσης από το κυβερνών κόμμα να ελευθερώσει όλους τους πολιτικούς κρατούμενους και να μπει σε διάλογο προκειμένου να βρεθεί πολιτική λύση. Ευχαριστώ πολύ κύριε Γκέρνγκερ. Ο κύριος Μιγκάλσκι για διαδικαστικό θέμα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Μα είπατε ότι η διαδικασία Catch the Eye θα καλύψει μόνο δύο ομιλητές. δεν θα αφήσετε αυτούς οι οποίοι μίλησαν στην προηγούμενη συζήτηση να λάβουν το λόγο στην τρέχουσα συζήτηση. Μα γιατί? Κάποιος ο οποίος μίλησε στην προηγούμενη συζήτηση δεν θα πρέπει να τύχει διακρίσεων επειδή θέλει να συμμετάσχει και στην τρέχουσα συζήτηση. Ίσως θα μπορούσατε να διευρύνετε λοιπόν τον κατάλογο των ομιλητών στη διαδικασία ΚΑΤΣΔΙ. Κύριε Μιγκάλσκι, κάνω ό,τι μπορώ αλλά υπάρχουν ορισμένα κριτήρια τα οποία θα πρέπει να τηρήσω σε σχέση με τη διαδικασία κατστιά, γιατί ακριβώς αυτή η διαδικασία έχει σαν στόχο αυτοί οι οποίοι δεν έχουν τη δυνατότητα από τις ομάδες τους να λάβουν το λόγο να μπορέσουν να συμμετάσχουν και αυτοί στη συζήτηση. Αυτό δεν οδηγεί σε κάποια διάκριση. Απλώς δίνει τη δυνατότητα στους συναδέλφους που δεν έχουν λάβει το λόγο προηγουμένως να μιλήσουμε πριν από αυτούς οι οποίοι θέλουν για δεύτερη φορά να λάβουν το λόγο. Και είχα μονάχα δύο λεπτά, έδωσα το λόγο σε τρεις συναδέλφους. Δεν μπορούμε λοιπόν να κάνουμε μια συζήτηση για το θέμα αυτό. Έχει κλείσει η συζήτηση και έρχομαι. Κύριε Μιγκάλσκι, δεν θα κάνουμε συζήτηση για αυτό το θέμα τώρα. Δίνω το λόγο στον Επίτροπο κύριο Κέλλας. Πρόεδρε, αξιότιμοι ευρωβουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ελπίζω να εγκριθεί το ψήφισμα του Κοινοβουλίου. Σημεριζόμαστε τις ανησυχίες σας για τις πρόσφατες εξελίξεις εκεί. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έδρασε από την αρχή, από τις εκλογές και καταδίκασε όλες τις βίες πράξεις που έλαβαν χώρα και ζήτησε από όλες τις πλευρές να συμμετάσχουν σε διάλογο για να διασφαλιστεί η διεξαγωγή ελεύθερων εκλογών. Δεν πήγε δεν πήγαν παρατηρητέ ε, λόγω της επικίνδυνης κατάστασης εκεί και πρέπει εδώ να αναφερθώ στο γεγονός ότι η Κάθριν Άστον συναντήθηκε πρόσφατα με τον Πρωθυπουργό του Μπαγκλαντές. Η βία οδήγησε σε πολλούς θανάτους και σε πολλούς τραυματισμούς. Τα θύματα περιλαμβάνουν και γυναίκες και παιδιά, αλλά και θρησκευτικές και εθνικές μειονότητες. Δυστυχώς, τα κύρια πολιτικά κόμματα απέτυχαν να συμφωνήσουν για τις προϋποθέσεις προκειμένου να διεξαχθούν εκλογές όπου να συμμετέχουν όλοι. Το κόμμα της αντιπολίτευσης, το BNP, εμποϊκόταρε τις εκλογές. Παρ' όλα αυτά έγιναν οι εκλογές. Κάτω από αυτές τις συνθήκες λοιπόν η αποστολή παρατηρητών δεν θα βοηθούσε. Ευχαριστώ πολύ πάντως για την ε, συνεργασία μέχρι τώρα. Πρέπει να ξέρετε ότι οι εκλογές, όπως είπατε κι εσείς, χαρακτηρίστηκαν από βία και η συμμετοχή ήταν χαμηλή. Τώρα λοιπόν ζητάμε να σταματήσει αμέσως η βία και επαναλαμβάνω και την έκκλησή μας για διάλογο. Ζητάμε από τους ε, ηγέτες και του κόμματος του κυβερνητικού και της αντιπολίτευσης να βρουν έναν τρόπο για να προχωρήσουν προς τα μπρος και να οργανώσουν αξιόπιστες εκλογές, να δώσουν σημασία στους πολίτες πρώτα απ' όλα, ώστε να υπάρξει μια δημοκρατική διαδικασία και έτσι τον Μπαγκλαντές να μπορέσει να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις, τις οικονομικές και κοινωνικές που έχει μπροστά του. Όπως επίσης και προκλήσεις σχετικά με την ασφάλεια των εργοστασίων και τις κοινωνικές συνθήκες. Εμείς θα συνεχίσουμε να βοηθάμε. Θα συνεχίσουμε να ελέγχουμε από κοντά την κατάσταση όσον αφορά τα ανθρώπινα και τα θεμελιώδη δικαιώματα και θα στηρίζουμε την δημοκρατική διαδικασία στον Μπαγκλαντές. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Κάλλας. Για τη λήξη της συζήτησης υπάρχουν έξι ψηφίσματα που έχουν κατατεθεί. Κλείνει η συζήτηση και η ψηφοφορία θα γίνει μετά την επόμενη συζήτηση. Επόμενο σημείο έχουμε των ε, μέτρων για την ποινικοποίηση των ΛΟΑΔΜ. Καταρχήν οι συντάκτες του ψηφίσματος